Οπότε υπάρχουν όμως ακόμα πολλά εμπόδια όπως γνωρίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να βοηθήσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Φεγγερέιντο παρακαλώ.